guten Tag. Wir sind in einem riesengroßen Raum. Καλημέρα σας. Θα ήταν καλό να ήμασταν όλοι έτοιμοι και όλοι παρόντες, αλλά δεν είμαστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που κάποιοι τουλάχιστον συνάδελφοι έχουν έρθει. Δεν φαίνεται πολύ γεμάτη η ημερησία διάταξη, αλλά έχει αρκετά πράγματα, μπορώ να σας πω. Να σας πω ότι γλώσσες έχει σήμερα στο πάλκο πάντα εκτός από σουηδικά, εστονικά, ε, λετονικά, λιθουανικά και μαλτέζικα. Όλες οι άλλες γλώσσες είναι στη διάθεσή σας. Είμαστε πάντα στο διαδίκτυο, στα ριάκια του διαδικτύου. Σας παρακαλώ λοιπόν να φέρεστε αντιστοίχω. ούτε να κοιμόσαστε, να διαβάζετε εφημερίδες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει κανείς στο διαδίκτυο, όταν βγαίνει στο διαδίκτυο προηγούμενη εβδομάδα μια μικρή αντιπροσωπεία πήγε στο Έσεν, στην πολιτιστική πρωτεύουσα, ο κύριο Στάκουλα και εγώ ήδη, ίδια και ορισμένοι ακόμα. Έχουμε μια έκθεση για την ε, επίσκεψη αυτή. Μπορώ να σας πω ήταν απλώς θαυμάσια αυτή η επίσκεψη. Είδαμε τις εκδηλώσεις για την πολιτιστική πρωτεύουσα και είδαμε πως υπήρχαν ουσιαστικά 53 ε, εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο ΕΣΕΝ. Ήταν μια πολύ καλή λοιπόν ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργεί ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Μάθαμε επίσης με την επίσκεψή μας στο ΕΣΕΝ, κάτι που ξέραμε ήδη από το Λουξεμβούργο και την επίσκεψη στο Ζάρλαντ και όπως ισχύει και στο Λίβερπουλ, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα παλιά εργοστάσια, τους παλιούς βιομηχανικούς χώρους για να τους χρησιμοποιήσει. Βέβαια υπήρχε και μια πολύ ωραία αίθουσα όπερας και είπε ο κύριος Στάκουλα τι ωραία που ένας Φιλανδός αρχιτέκτονας είχε φτιάξει αυτό το κτίριο της όπερας στο Έσεν. Εμείς δεν μπήκαμε μέσα, το είδαμε μοναχα απ' έξω το κτίριο. Αλλά οι πολιτιστικοί χώροι που είδαμε, το νέο μουσείο του Ρουρ, όλα αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα του πώς μπορούν να αναζωογονηθούν οι χώροι, οι παλιοί βιομηχανικοί χώροι, ώστε και στο μέλλον να μπορέσουν να παίξουν ένα ρόλο πολιτιστικό για τα παιδιά και τα εγγόνια μας που ποτέ δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν με τα μάτια τους πώς λειτουργεί ένα ορυχείο παραγωγής χάρη, αλλά μπορούν θαυμάσια να δουν με αυτούς τους χώρους πώς ήταν στο παρελθόν τα πράγματα. Στους χώρους αυτούς μπορούν να χρησιμοποιούνται και για πολιτιστικά γεγονότα. Θα έχετε την έκθεση στην ε, έκθεσή σας. Η Κωνσταντζ νομίζω ότι έχει κάνει μια πολλή έκθεση. Και τώρα η τελευταία μου παρατήρηση. Θέλω να σας πενθυμίσω, δυστυχώς, σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση, μια στρογγυλή τράπεζα, πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης, εξωτερικές σχέσεις στις 6.30 μέχρι τις ε, 8,5, 9, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν κάποιοι από εσά προτιμούν να δούνε ποδόσφαιρο, εγώ προσωπικά θα πρέπει να μείνω. Ξέρω ότι παίζει και η χώρα μου. Είχαμε περίπου 60 άτομα τα οποία είχαν πει ότι θα έρθουν. Λοιπόν, κάντε μια προσπάθεια να έρθετε και ορισμένοι από τους συναδέλφους μας έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αναπτύξουν αυτή την εξωτερική διάσταση στα πολιτιστικά θέματα. Έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε και το θέμα του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Θα γίνει βέβαια μόνο στα αγγλικά αυτή η εκδήλωση. Δεν ήθελα να έχουμε μια τέτοια συνεδριάσεων. Να έχουμε ένα μικρό όμως και πιο ε, άνετο χώρο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας κανονικά. είμαστε τώρα στο κανονικό μας, στα κανονικά μας θέματα, στη μέρησια διάταξη. Έχουμε σήμερα την ψηφοφορία για τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωση, τη δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη. Ο Μόρτεν Λόκεγκαρτ είναι ο εισηγητής. Έχουμε καμία διακόσαριά περίπου τροπολογίες, αλλά έχουμε και τις συμβαστικές τροπολογίες του εισηγητή. Μπορούμε να ψηφίσουμε με ανάταση χειρών. Τώρα, αν δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε την ε, κάρτα, όχι την πιστοτική, την κάρτα ψηφοφορία. Αν θέλετε, βάλτε την ήδη στην απαραίτητη σχισμή για να είστε έτοιμοι, να χρειαστεί να ψηφίσουμε. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Λόκεγκαρτ, το λόγο για να μα παρουσιάσει την εκθεσή του με λίγα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουν υποθεί ήδη αρκετά για αυτήν ε, την έκθεση, οπότε δεν θα παρατείνω τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απλώς μερικούς ε, συναδέλφους, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην έκθεση αυτή. Ειδικότερα τους κοιόδες εισηγητές για τη συμβολή του, τη συμμετοχή του στην όλη διαδικασία. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συναντήσεις και συζητήσεις επί τη βάση των ε, πολλών τροπολογιών σας. Να ευχαριστήσω επίσης ε, την Επιτροπή, του εκπροσώπους της ε, Επιτροπής για μια επικοδομητική και ανοιχτόμυαλη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να το περιμένουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ επικοδομητικέ οι συζητήσει και με του εκπροσώπου τη Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίση τη γραμματεία τη Επιτροπή μα ε, για τα πρακτικά αλλά βέβαια και στους βοηθούς μου για την υποστήριξη και τη σκληρή δουλειά τους καθ' όλη τη ε, διαδικασία αυτή. Ελπίζω οι προσπάθειες αυτές να αντικατοπτριστούν στη σημερινή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα ακολουθήσει η συζήτηση. Η συζήτηση έχει γίνει και απλώς θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας δώσω τώρα για περαιτέρω συζήτηση. Άμα θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση για τις τροπολογίες, όταν φτάσουμε εκεί θα ζητήσουμε. Περισσεύει ένας βουλευτής από το ΕΛΚ, νομίζω. Ποιος εθελοντικά δεν θα ψηφίσει. Ποιος. Εντάξει. Ωραία, πολύ, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, απλώς ήθελα να σας πληροφορήσω γι' αυτό. Περισσεύει και ένας από την ΚΟΕ. Κάποιος θα πρέπει να μην ψηφίσει, λοιπόν. Δεν θα συμμετάσχουν ο κύριος Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δύο ψήφους έχει το κόμμα σας, όχι τρεις. Ερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία. Παράγωγος 1, τροπολογία 32, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτήμα. Θα αναφέρω μονάχα τις τροπολογίες, δεν σας λέω τώρα παραγράφους. 33. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 καβαντά υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές, θέλουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφι υπέρ. Λοιπόν, ναι, ναι. κλείνω την ψηφοφορία, την ηλεκτρονική. Απέριπτε. 12-8. 8 υπέρ, 12 κατά δηλαδή. Μήπως μπορώ να πάρω ένα κατάλογο ψηφοφορίας από το ΕΛΚ. Λέει πρόεδρος. 36 ψήφοι υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ τα αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 47 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 47 Άρχεται. Ψηφοφορία. Πέρας. 11-11 απορρίπτεται. 48. Μάλιστα. Έχετε πρόβλημα με τη μηχανή σας. Δεν δουλεύει. Καθίστε πίσω Κύριε Μάτουλα, πηγαίνετε πίσω. Μπορείτε να βοηθήσετε τον συνάδελφο. Σαράντα ψήφι υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Πέρας. 16-12 γίνεται δεκτή. Πάντα πρέπει να τα κάνουμε όλα δύο φορές. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 59. Ψήφι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρα τούτε. 19-9 δεκτή. 60 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 62 υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. 63, 64 και 65 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτές. 66 έχει αποσυρθεί. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίβεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 <clears throat> και 81 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτει. 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ έχει εκπέσει λέει η γραμματεία. Εκπίπτει, εκπίπτει 83. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε στον 84. Ψήφι υπέρ στην 84. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 95 και 96 είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Η 97 εκπίπτει. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 99 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. I would like to withdraw this amendment. Αποσύρω αυτή την τροπολογία και θέλω να θέσω μια προφορική τροπολογία που τροποποιεί το πρώτο τμήμα αυτής της τροπολογίας. Λέγον, αναγνωρίζει τη σημασία των Euronews και τη σημασία του να επεκτείνει το γλωσσικό του φάσμα το Euronews για να καλύψει όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να είναι ένα υπόδειγμα τηλεοπτικής δημοσιογραφίας που θα δώσει μια πληροφόρηση η οποία θα είναι μεγάλης ποιότητας και θα έχει και την διαφάνεια και τις διαφημίσεις που απαιτούνται. Το κατάλαβα, αλλά ίσω όχι, δεν έχουν, έχουμε άλλο το κείμενο εγώ, αλλά κανένα άλλο δεν έχει. Το ξαναδιαβάζω, λέει η πρόεδρο. Αν κάποιο ε, έχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Το ξαναδιαβάζω. Αναγνωρίζει τη σημασία των Euronews, τη επέκταση μάλλον από την πλευρά του Euronews, του γλωσσικού φάσματο για να καλύψει όλα τα κρατη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επέκεινα και επίσης του να είναι το Euronews ένα υπόδειγμα ανεξάρτητο, ανεξάρτητης τηλεοπτικής δημοσιογραφίας που προωθεί την αντικειμενικότητα στην πληροφορία, την ποιότητα στην ε, πολιτική και την διαφάνεια στις διαφημίσεις. Κοιτάξτε, δεν, δεν έχω πρόβλημα. Well, just, uh, <laughs> just thinking of the text. Uh, Εντάξει, σκέφτομαι λίγο και το κείμενο. Το, αυτό που συζητούμε τώρα είναι αν πρέπει να υποβληθεί ή όχι και όχι το κείμενο αυτό καθ' αυτό. Εντάξει τότε. Okay. Yeah. Κύριε Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένα απλό σχόλιο στη συνάδελφο που μόλις κατέθεσε αυτή την προφορική τροπολογία. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το Euronews θα μπορούσε να γίνει, θα γινόταν ανεξάρτητη, ανεξάρτητος τηλεοπτικός σταθμός. Είναι. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ε, θα εξακολουθεί να είναι. Μπορούμε να δεχτούμε αυτή την αλλαγή. Δέχεται η κυρία Παλιαδέλη. Thank you. Um, Ζητήσαμε χωριστή ψηφοφορία. Τώρα με την προφορική αυτή τροπολογία δεν χρειαζόμαστε πια χωριστή ψήφο. Μπορούμε να ψηφίσουμε ολόκληρη την τροπολογία. Ψηφίσουμε την τροπολογία της κυρίας Παλιαδέλη όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Κάβαντα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 100. Υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Δεκτή. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 103, 104 ταυτίζονται ψήφι υπέρ κατά απόχέ εγκρίνονται. 105 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται. 106 και 107 είναι ταυτόσιμε υπέρ κατά αποχέ δεκτέ. 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα 112, 13 μέχρι 120 έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Ποιος είναι υπέρ των τροπολογιών 111 112 έως 120. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Είναι τροπολογίες της διαγραφής του ή 121. Εκπίπτει 121 και η 122 επίσης. 123 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. <clears throat> Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 124 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία για την 124. Πέρας. 17-10 γίνεται δεκτή. Τρο, προφορική τροπολογία του κυρίου Μπέλετ. Υπαριθμόν 1. Πρέπει να το εξηγήσετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχετε το κείμενο. Θαυμάσει. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 125. Εκπίπτει, εκπίπτει, ναι, ναι. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1-3-2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 133. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 139 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 2 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 142 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά έλεγχος 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 11-18 απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 146, 147 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. 148 υπέρ, κατά, πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 148. Πέρας. 15-15 απορρίπτεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 158. Πέρας. 13-15 απορρίπτεται. 159 και 160 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165, 66 και 67 ταυτόσιμες ψηφί υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβαστική 8 <clears throat> ψηφί υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 15-15 απορρίπτεται. 169 και 170 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτονται. 171 απερίφ, απεσύρθη, 172 ψήφι υπέρ. Κατά, απόχέ απορρίπτονται. 173 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες από κοινού. 174 μέχρι 185. Όχι, δεν μπορούμε. Καλά, αφού δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. 174. 174. Ψήφι υπέρ. Κατά έλεγχος. 174 έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Δεκτή. 17-13. 176 υπέρ. Δεν θέλετε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Τι να κάνω. Υπέρ 176. Έλα, στα γρήγορα. Κατά. χες Λοιπόν, Πάλι σηκώστε τα χέρια. 176 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Πάλι έλεγχο χρειάζεται. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ε, άρχεται ηλεκτρονική, λίγη ηλεκτρονική. 18-11 εγκρίνεται. Ωραία. Κύριε Καβαλά. Ναι, κυρία Πρόεδρε από την 75 μέχρι την 95 να τις ψηφίσουμε unblock από την 175 μέχρι την 185 μπορούμε να τις ψηφίσουμε unblock. Η κυρία Βερζέ είπε 9. Δεν μπορεί να ψηφιστεί. Τι να κάνουμε. 175 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 181 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 185 κατά αποχές 185 υπέρ κατά αποχές δεκτή ένταξη 1 υπέρ τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε <clears throat> για την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 15-15 απορρίπτεται. 8 ψήφι κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 και 12 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 20 υπέρ, κατά. Πρέπει να ελέγξουμε για την 20. Αυτή την ψηφοφορία. Πέρας. 25 25-5. Θα φαινο, φαινότανε. Άλλη φορά, άλλη φορά να μην κάνουμε αυτή τη γυμναστική. Πρέπει να κάνουμε αεροβική εδώ πέρα με τα χέρια μας, μια φορά το δεξί, μια φορά το αριστερό χέρι και τελειώνει. 21 και 22 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτονται. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25. Μήπως μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι τον 25 με 31 όλες μαζί. Εντάξει. 25 μέχρι 31. Ψήφι υπέρ κατά αποχές περάσαμε. Τελική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ ηλεκτρονικά με την κάρτα σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Λόκεγκαρτ. Ωραία. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερησής διάταξης. Είναι το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η κυρία Παλιαδέλη είναι η συγγήτρια. είναι η συγκεντριά μας για την έκθεση αυτή. Είχαμε την τελευταία φορά την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων για το ζήτημα αυτό. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε τα κείμενα αυτά από τα εθνικά κοινοβούλια. Και ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε η Γαλλική Γερουσία για αυτό το ευρωπαϊκό σήμα. Αξίζει το, να το διαβάσετε. Οι Γερμανοί ήταν υπέρ, οι Γάλλοι ήταν κάπως διηρημένοι σε αυτά τα θέματα, αλλά ήταν χρήσιμο να δείτε τι λένε τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια για το θέμα αυτό, γιατί είναι επιχειρήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση. Κυρία Παλιαδέλη, σα δίνω λοιπόν το λόγο για να μα παρουσιάσετε τη θέση σα για αυτό το σήμα Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρομία. Ότι η άρνηση γαλλική γερουσία δεν είχε σχέση νομίζω με την ουσία, είχε σχέση με την ουσία του ζητήματος για το αν δηλαδή έχει μια προστιθέμενη αξία το σήμα της πολιτικής κληρονομιά, ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι με τις απαντήσεις που περιμέναμε από τα κοινοβούλια τα οποία καλούνται να διευκρινίσουν αν εμπίπτει στην αρχή της επικουρικότητας ή όχι. Δηλαδή άλλη δουλειά των κοινοβουλίων και άλλη απάντηση της Γερουσίας αυτή την εντύπωση έχω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι με τιμά ιδιαίτερα ότι η Επιτροπή Πολιτισμού μου εμπιστεύτηκε να εισηγηθώ την πρόταση για την κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να ομολογήσω ταυτόχρονα ότι θεωρώ μεγάλη ευθύνη όχι, το, τη θεωρώ μεγάλη ευθύνη αυτή την έκθεση, όχι μόνο επειδή αναφέρεται σε μια δράση που θα προκύψει με συναπόφαση, αλλά κυρίως επειδή αφορά σε ένα θεσμό που στοχεύει στην ενίσχυση της αίσθησης των Ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει κοινών στοιχείων ιστορίας και κληρονομιάς. Κεντρική ιδέα του σήματος είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά ως εργαλείο για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας αφορά σε χώρους των κρατών μελών που είτε σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό, είτε με την οικοδόμηση της Ενωμένης Ευρώπης. Η αρχική ιδέα διατυπώθηκε το 2005 από τους Υπουργούς Πολιτισμού των κρατών μελών ως μία από τις απαντήσεις στο έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της και ενώ που συσχετίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την έλλειψη γνώσεων, έτσι τουλάχιστον εκτιμήθηκε, για την ιστορία της Ευρώπης, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες στις οποίες αυτή βασίζεται. Εκτιμώ βεβαίω ότι η διαπίστωση αυτή δεν ανταποκρίνεται απολύτω στην πρόσφατη τουλάχιστον πραγματικότητα και δεν βαρύνει επομένω του Ευρωπαίου η έλλειψη κοινωνική συνοχή, αλλά κυρίω του ηγέτε του που βρέθηκαν απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα οικονομική κρίση ή να υπερβούν τα όρια των εθνικών κρατών. Από τη στιγμή όμως που θεωρείται ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε μέσα από, την, από τον πολιτισμό προκειμένου να πετύχουμε την κοινωνική συνοχή, το δέχομαι και συνεχίζω. Από το 2006 ο θεσμός υλοποιήθηκε σε διακυβερνητικό επίπεδο με τη συμμετοχή 17 ευρωπαϊκών κρατών, ανάμεσά τους και την Ελβετία, και 64 συνολικά χώρους να γίνονται αποδέκτες του σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς τον Νοέμβριο του 2008 τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να μετατρέψει τη διακυβερνητική πρωτοβουλία σε επίσημη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομιλούσα ανέλαβε την ευθύνη να εισηγηθεί για την πρόταση συναπόφαση της 22 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Η ίδια και οι συνεργάτες της συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της Κομισιόν, του Συμβουλίου, της Επιτροπής Περιφερειών, μέλη της Ευρώπα Νόστρα, οργανώσεις τη Κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, και συζητήσαμε με ειδικού για το περιεχόμενο του σήματο και τι διαδικασίε απονομή του. Ιδιαίτερα επικοδομητική υπήρξε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων τη εισηγήτριας με του σκιώδει εισηγητές στις 16 Ιουνίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε σημαντική σύμπτωση απόψεων σε ό,τι αφορά στον ορισμό των αποδεκτών του σήματο, την αποσαφήνιση των κριτηρίων και άλλα στοιχεία. Διάχυτη κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτή ανταλλαγή απόψεων, κυρίω όμως η διάθεση για δραστικέ παρεμβάσει στην ουσία και όχι μόνο στο κείμενο τη πρόταση ήταν από τα στοιχεία που διαπιστώσαμε στην, κατά τη συζήτηση με τους σκιώδει συζητητέ. Πιο συγκεκριμένα, ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι αν η δράση θα περιοριστεί, σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στα 27 κράτη-μέλη, όπως προτείνεται στο άρθρο 4, ή αν θα υπερβεί τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δηλαδή θα παραμείνουμε στους 27 για τους 27 ή αν θα υπερβούμε τα όρια της Ένωσης και θα γίνουμε περισσότεροι. Κατά την εκτίμησή μου και με δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά υπερβαίνει τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σήμα θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να πονέμεται σε μνημεία, τόπους, ιδέες που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στη γεωγραφική διάσταση της Υπήρου. Στην Ευρώπη δηλαδή και τα κράτη που την αποτελούν, άσχετο αν είναι ή δεν είναι μέλη της. Το γεγονός ότι οι μνημεία στην Ελβετία έχουν ήδη λάβει το σήμα, όταν ακόμη το σήμα ήταν διακυβερνητικού χαρακτήρα, αποδεικνύει την ανάγκη για τη διεύρυνση του θεσμού εντό των ορίων τη Ευρώπη και όχι τον περιορισμό του στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια επιλογή θα προσέδιδε στο σήμα μια ακόμη μεγαλύτερη συμβολική προστιθέμενη αξία. Δεδομένη μάλιστα τη μελλοντική επέκταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το σήμα θα λειτουργούσε θετικά στη διαδικασία ένταξη. Το ενδεχόμενο μάλιστα το σήμα να αποτελέσει απόδοση Uh, το ενδεχόμενο μάλιστα το σήμα να αποτελέσει απόδοση τιμής σε θέσεις εκτός Ευρώπης που εμπίπτουν στα κριτήρια επιλογής, ανεβάζοντας έτσι το πολιτιστικό πρεστής της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια ιδέα που έπεσε από έναν συνάδελφο Σκιώδη, ε, θα ήταν μια πολύ φιλόδοξη προοπτική που δεν θα έπρεπε να την αποκλείσουμε εκ των προτέρων. Αυτό που πιστεύω στο σημείο αυτό είναι ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Υπήρου θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποψηφιότητα για την απονομή του σήματος αυτού, εφόσον εκτιμά ότι πληρεί τα κριτήρια. Σημαντικό ζήτημα για το, για κύρος του σήματος και τη διαφάνεια στην απονομή του αποτελεί η σαφής διατύπωση των κριτηρίων του στο άρθρο 7, προκειμένου να αποφευθούν ασάφειες ή παρατυπίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της δράσης σε διακυβερνητικό επίπεδο. Σύμφωνα με την πρόταση, οι χώροι πρέπει να ανταποκρίνονται στη σχέση τους με την, ε, με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης που εφόσον είναι πολιτισμική θα έλεγα μπορεί να περιλαμβάνει και μνημεία όπως για παράδειγμα τα μουσουλμανικά της Ιβηρικής Χερσονήσου που δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκά με την ε, τρέχουσα σημασία του όρου. Δεύτερον, στη συμβολή του στην οικοδόμηση της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι εντελώς σαφές, περισσότερο προς το δεύτερο. Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη ως ιδέα ανάγεται σε χρόνια πολύ παλαιότερα βέβαια, στον Καρλομάγνο τουλάχιστον αν όχι και παλιότερα, αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σαφή ημερομηνία γέννηση. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σήμα έχει δύο σαφώς, έτσι όπως ορίζεται στην, στην απόφαση, έχει δύο σαφώς διακριτά σκέλη, πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και ε, η Ενωμένη Ευρώπη, που θα πρέπει να μας αποσχολήσουν και στο επίπεδο των κριτηρίων αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το κύρος του. Ο προπολογισμό του άρθρου 14 είναι ένα ζήτημα που μα απασχόλησε, επειδή είναι και κλειδί αλλά και αγκάθι για μια πρωτοβουλία δράση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κονδύλιο που θα διατεθεί με βάση την πρόταση είναι περί το 1.350.000 ευρώ και αφορά στα λειτουργικά έξοδα εφαρμογή τη δράση για μία τριετία, δηλαδή τη γραμματιακή υποστήριξη και τις δαπάνες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και την περιορισμένη υποστήριξη δράσεων στους βραβευμένους χώρου. Από την άποψη αυτή το σήμα δεν αποτελεί αφορμή για χρηματοδότηση, για υποδομές ή καλλιτεχνικές δράσεις όπως της πολιτιστική πρωτεύουσα ο θεσμός, αλλά για επιβράβευση χώρων που καλύπτουν με την κατάθεση της υποψηφιότητά τους τα κριτήρια που απαιτεί η απονομή του σήματος. Δηλαδή ένα ένας χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για να, προκειμένου να λάβει το σήμα. Εκτιμώ ωστόσο ότι μια βράβευση με χρηματικό σκέλος θα συνέβαλε στην προστιθέμενη αξία της κοινοτική δράσης σε σχέση με τη διακυβερνητική φάση της, εφόσον, και αυτό θα μπορούσε να γίνει εφόσον μειωνόταν ο αριθμός των τελικών αποδεκτών του σήματος, όπως προτείνουμε στη συνέχεια. Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα είναι στο άρθρο 10 και 11, όπου προτείνεται, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, κάθε κράτος να υποβάλει ετησίως δύο υπό, ε, υπό ε, έγκριση ε, χώρους. Επομένως, 54 συνολικά προτάσεις, από τις οποίες θα επιλέγονται ετησίως δυνητικά όμως 27, μία αναχώρα. Αυτό σημαίνει ότι στα τρία πρώτα χρόνια εφαρμογής της δράσης είναι δυνατό, όχι αναγκαστικά ότι έτσι θα γίνει, να λαμβάνουν το σήμα 81 χώροι στα τρία χρόνια της πρώτης εφαρμογής. Μια τέτοια λογική εκτιμώ ότι αφαιρεί από το κύρος του σήματος, ανάγει την όλη διαδικασία σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα χωρίς προστιθέμενη αξία και κυρίως μεγιστοποιεί τη λειτουργική δαπάνη, ακυρώνοντας τη δυνατότητα για παράλληλη με την απονομή χρηματοδότηση των αποδεκτών του σήματος. Θεωρώ ότι αν μειωνόταν δραστικά ο ετήσιο αριθμό των αποδεκτών, το σήμα Ευρωπαϊκή Πολιτική Κληρονομιά θα γινόταν μια πραγματική απόδοση τιμή σε θέσεις που πραγματικά θα ανταποκρίνονται στα κριτήρια επιλογής για τη συγκεκριμένη δράση. Ένα άλλο ζήτημα μικρότερης σημασίας είναι η αιτήσια ή η διετής ενεργοποίηση της δράσης. Αν μειωθεί δραστικά ο αριθμός των αποδεκτών, η απονομή μπορεί να είναι αιτήσια. Αν όμως διατηρηθεί ο σημερινός αριθμός, ο δυνητικός δηλαδή των 21 κάθε χρο... των 27 κάθε χρονιά, ε, θα πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση. Παραδείγματος χάρη μια αναδιετή απονομή ένα ένας θεματικός ανακατηγορία και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τους εμπειρογνώμονες, την ομάδα δηλαδή που θα απαρτήσει αυτούς που θα επιλέξουν ε, ε, ε, τους χώρους που θα βραβευθούν, ε, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8, ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, διαφυλάξουμε τη διαφάνεια και τη σοβαρότητα της δράσης. Επομένως, οι εμπειρογνώμονες πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να το κάνουν. Με την παρούσα πρόταση προτείνονται 12 ε, συνολικά μέλη σε αυτή την πρόταση, ε, όπου 4 είναι από το Κοινοβούλιο, 4 από την Κομισιόν και 4 από το Συμβούλιο. Ε, θεωρώ ότι ο ζυγός αριθμός των μελών θα πρέπει να γίνει μονός. Επομένως, θα μπορούσε να είναι ένας εκπρόσωπος που θα οριζόταν από την Επιτροπή των Περιφερειών, για να έχουμε ένα αριθμό 13 ε, ε, μελών στην ομάδα αυτή των εμπειρογνώμων. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ειδικοί αυτοί θα πρέπει να, είναι, ε, να, να έχουν ειδικότητα σε περισσότερα από ένα θέματα, να γνωρίζουν την ευρωπαϊκή ιστορία, να μπορούν να, διαχειριστούν, να, να, να κατανοούν τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών κλπ. Και βέβαια καλά θα ήταν η εκπροσώπηση αυτή ε, να μην περιορίζεται στους τρεις θεσμικούς φορείς, την Κομισιόν, την την, το Συμβούλιο και την, το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά να είναι και γεωγραφικά ισορροπημένη. Σε ό,τι αφορά την τελική επιλογή, όπως περιγράφεται στα άρθρα 11 και 13, το πάνελ των εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις υποψηφιότητες και συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει σύσταση για την απονομή του σήματος. Η τελική επιλογή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Επιτροπή. Βασίζεται όμως στην έκθεση του πάνελ, του, του, του πάνελ των εμπειρογνωμόνων. Ε, θα πρέπει να γίνει σαφέ, με ανησύχησε λιγάκι, η αυξημένη αυτή αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία από τη διατύπωση στην, στην αρχική πρόταση μια, μοιάζει να μην δεσμεύεται απολύτω από την απόφαση τη ομάδα των εμπειρογνωμών. Σε μια επαφή όμω με, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πήρα τη διαβεβαίωση ότι στην πράξη δεν θα επανεξετάζει τι υποψηφιότητε, απλώ κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθεί την πρόταση τη ομάδα. Ε, θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε ίσω τρόπου με του οποίου θα, μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ αυτή την κατεύθυνση, προ την απονομή δηλαδή. Να μετέχει, να συμβάλλει, να επικυρώνει. Ακόμη δεν το έχω βρει, δεν ξέρω αν νομικά επιτρέπεται, θα το ψάξουμε. Ε, το επόμενο θέμα αναφέρεται στο άρθρο 12 και αφορά στου διακρατικού χώρου, τα transnational ε, ε, areas. στου χώρου δηλαδή που αφορούν περισσότερο από ένα κράτη-μέλη. Ε, προτείνουμε σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής ότι δεν ε, υποβάλλει ένα μονοκράτος μέλος αλλά πρέπει να συμφωνήσει και ένα άλλο κράτος μέλος προκειμένου να κατεβάσουν κοινή πρόταση που να αφορά το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος αν έχει δύο δυνατότητες προτάσεων τη μία θα τη χάσει επειδή θα προτείνει μια, έναν χώρο μαζί με κάποιο άλλο μέλος ε, με το οποίο έχει κιόλα συμφωνήσει να συνυποβάλλουν την υποψηφιότητα. Υπάρχει ένα ζήτημα μεταβατικών διατάξεων στο άρθρο 18 που ε, αφορά στο αν θα διατηρήσουμε ή θα επιστραφεί ή τι θα γίνει τέλος πάντων με το διακυβερνητικό σήμα. Δηλαδή με αυτές τις θέσεις που ήδη έχουν πάρει το σήμα στην προηγούμενη φάση. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαχωρίσουμε τα δύο σήματα και ως προς τη μορφή και ως προς τη διαδικασία απονομής. Οι χώροι που το έχουν λάβει, το προτείνω αλλά είμαι ανοιχτή σε άλλες προτάσεις, θα πρέπει να διατηρήσουν το παλιό και εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια της νέας φάσης, της προκήρυξης δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποβάλουν εξ αρχής πρόταση προκειμένου να του απονεμηθεί εφόσον πληρούν τα κριτήρια. Ε, και ένα τελευταίο ζήτημα που αφορά στο λογότυπο, κάτι που δεν θίγεται στην πρόταση, πρέπει να προσθεθεί. Εκτιμώ ότι για τη διαφοροποίηση του σήματο από το διακυβερνητικό παρελθόν του θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο λογότυπο μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, κάτι που εκτιμώ πως θα διευκόλυνε το ζήτημα τη διατήρηση ή όχι του σήματο τη διακυβερνητική πρωτοβουλία. Τελειώνοντα, θέλω να επισημάνω τα ακόλουτα. Η πρόταση της Κομισιόν παρά τις πολύ καλές της προθέσεις, έχει χαρακτηριστικά γραφειοκρατικής προσέγγισης, που αντιμετωπίζουν διστακτικά και ας μου επιτραπεί χωρίς όραμα έναν θεσμό που θα έπρεπε να αξιοποιηθεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός της Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, εξακολουθεί να είναι ίσως το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Υπήρου μας ως εργαλείο, δηλαδή θα έπρεπε να το δούμε αυτό το σήμα, ως εργαλείο κοινωνικής σύγκλησης και πολιτιστικής διείσδυσης και όχι ως έκφραση μιας λογιστικής, λογικής ισομοιρίας που νομίζω πως εν τέλει θα επηρεάσει αρνητικά το κύρος του θεσμού αλλά και την βιωσιμότητά του στο μέλλον. Αυτό όμω είναι μια προσωπική άποψη. Απλώ θεώρησα τον εαυτό μου υποχρεωμένο να την καταθέσω σε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και λίγο σκληρή, είμαι ανοιχτή στην αναθεώρηση, αλλά σταματώ εδώ, περιμένω τις δικές σας απόψεις, με την ελπίδα πως θα συμβάλλουν προσυστικά στη σύνταξη του σχεδίου έκθεσης που θα καταθέσω στο τέλος, στα μέσα του επόμενου μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σάντσε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα για την ανταλλαγή απόψεων και ακούγοντας ε, την εισηγήτρια την κυρία Παγιαδέλη, είπαμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί είναι ένα ζήτημα που φαίνεται αρκετά ευρύ και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε ό,τι θέλουμε σε αυτή την έννοια. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η ευρωπαϊκή κληρονομιά. Είναι μια πολιτιστική πτυχή, όπως ε, μόλις είπε η κυρία Παλιαδέλη, μήπω υπάρχει και μια ιστορική διάσταση επίσης. Είναι η αίσθηση του να ανήκει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που νομίζω ότι θέτουν κάποια ερωτήματα. Μιλήσατε για μνημεία πολλέ φορές. Δεν νομίζω όμως ότι αφορά μόνο μνημεία, αφορά χώρου ενδεχομένω και άειλη κληρονομιά. Όταν ε, βλέπουμε τους χώρους που έλαβαν αυτό το σήμα, δεν είναι μόνο μνημεία. Και το ερώτημα, το βασικό, είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του σήματος. Τι θέλουμε να επιτύχουμε ο προπολογισμό ε, τι θα επιφέρει στις συγκεκριμένους χώρους. Είναι θέμα επικοινωνία, ε, θα υπάρξει μια δικτύωση, υπάρχει μια τουριστική πτυχή, όπως, συμβαίνει στην περίπτωση του σήματος της UNESCO ας πούμε. Και ποιο είναι ο αριθμός των χώρων. Θέλουμε 27 κατέτος αν θέλουμε να βασιστούμε στο ότι το σπάνιο ε, είναι το καλύτερο, μήπως θα έπρεπε να είναι και λιγότερο, λιγότερα από 27. Ίσως να μην έπρεπε να είναι μόνο μνημείο, να μπορεί να είναι μία δράση, να μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Και ποιος θα είναι ο δικός μας ρόλος ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει και ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την απόφασή τη. Γιατί να μην εμπνευστούμε από τη διαδικασία που ακολουθείται για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Μου φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετέχει και είναι καλύτερα. Όχι, κάνω λάθος. Το σημείωμα νομίζω που έλαβα εγώ αναφέρεται σε μία γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα να εκφέρουμε κι εμείς την άποψή μας. Και τέλος, τι θα ζητήσουμε από τις χώρες για να είναι υποψήφιες. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια δέσμευση των ε, κρατών μελών, αλλά γιατί ακριβώς δεσμεύονται και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Τι προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να μπορέσει κανείς να λάβει το ε, ευρωπαϊκό αυτό σήμα. Θα είναι διαφορετικές οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθενται κατά με. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε φυσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ιδέα μου φαίνεται πολύ καλή, αλλά έχω να κάνω και κάποια ερωτήματα. Κάποια από αυτά καλύφθηκαν ήδη από την προλαλή σας, την κυρία Σάντσεφ Σμιτ. Το πρώτο μου ερώτημα είναι ότι εγώ από ό,τι κατάλαβα έχουμε μια πρόταση δύο ε, χώρων, δύο οντοτήτων κατά κράτος. Αλλά δεν ξέρω με κάθε σεβασμό τώρα μια χώρα όπως η Μάλτα δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αριθμό χώρων όπως η Γερμανία. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο μεγάλες και γι' αυτό έχουν μεγαλύτερη πολιτιστική κληρονομιά από ό,τι μικρές χώρες. Γι' αυτό μου φαίνεται κάπως παράξενη διατύπωση δύο χώροι για κάθε κράτος. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για προτάσεις που γίνονται από τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προτείνει κανείς τέτοιους χώρους, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οι ενώσεις πολιτών να μπορέσουν να διατυπώσουν προτάσεις αυτού του είδους. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα αυτής της ύπαρξης η οποία θα εξετάσει τις υποψηφιότητες θα ήθελα όμως να ξέρω ποιος παίρνει την τελική απόφαση, η Κομισιόν και μόνο ή θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει κάποιο λόγο στο θέμα αυτό. Και μετά υπάρχει και μια υποχρέωση να συντηρηθούν αυτοί οι χώροι. <clears throat> Τι ακριβώς προβλέπετε. Όχι μονάχα, δηλαδή να παρουσιαστεί μια υποψηφιότητα, θα πρέπει να υπάρχει και μια προστασία και συντήρηση των χώρων. Αν δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, θα αποσυρθεί το Ευρωπαϊκό Σήμα ή όχι. Ο κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχουν παρουσιάσει οι συνάδελφοί μας σε αυτό το χρονικό σημείο. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, κάπως, είναι αρκετά ικανοποιητικά. Ίσως μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα και στη συνέχεια. Αλλά εγώ θα είχα μια συζήτηση σε σχέση με την επιλογή των τόπων. Η επιλογή αυτών των τοποθεσιών θα πρέπει να γίνει από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Επομένως, θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σήμα για πολιτιστικού χαρακτήρα περιοχές. Αλλά αυτές οι περιοχές θα πρέπει να διατηρηθούν στο διηνεκές. Υπάρχει το άρθρο 14 το οποίο προβλέπει μια διαδικασία εποπτείας η οποία θα πρέπει να οδηγεί σε μια επικαιροποίηση κάθε τέσσερα χρόνια. Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να υπάρχει η εποπτεία αυτών των χώρων η οποία κοστίζει, θα κοστίζει περαιτέρω χρήμα. Και αυτό το οποίο με εκπλήσει είναι ότι όταν γίνει η επιλογή από τους ε, εμπειρογνώμονες, ενώ γίνεται από εμπειρογνώμους η επιλογή, τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία θα πρέπει να συντηρούν αυτούς τους τόπους, τις τοποθεσίες. Γι' αυτό εγώ προτείνω το εξής. Το κράτος μέλος, αντί για αυτή την υποχρέωση εποπτείας και επαλήθευσης κάθε τέσσερα χρόνια. Φυσικά το κρατός μέλος έχει κάθε συμφέρον να διατηρήσει αυτούς τους χώρους. Θα είναι καλύτερο το ίδιο το κράτος μέλος να κρατήσει λοιπόν σε καλή κατάσταση αυτούς τους χώρους. ή να μπορεί το ίδιο το κράτος μέλος να αποσύρει το ευρωπαϊκό σήμα όταν θεωρεί ότι δεν έχει νόημα η συντήρηση αυτού του χώρου. Επίσης και στην περίπτωση που έχει δοθεί αυτό το σήμα χρειάζεται μια αξιολόγηση εκ των υστέρων γιατί υπάρχουν πολλοί χώροι, πολλές τοποθεσίες που θα μπορούν να πάρουν αυτό το σήμα. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής αν ένας από αυτούς τους χώρους δεν εκπληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί στη συνέχεια να ξαναπροταθεί αυτός ο χώρος, αυτή η τοποθεσία. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τεθεί υποψηφιότητα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό εξαρτάται βέβαια από το αν είναι το κράτος μέλος το οποίο κάνει την επιλογή. Ελπίζω να με έχετε κατανοήσει και ελπίζω ότι κάθε φορά που ένα κράτος μέρος προτείνει μια τοποθεσία θα μπορεί να τίθεται υποψηφιότητα. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχουμε με αυτό το σήμα. Κύριο Σταβάρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις περιπτώσεις όπου <clears throat> στην πράξη έχουμε συμφωνήσει αλλά στο θεωρητικό επίπεδο ακόμα δεν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Δηλαδή συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το ευρωπαϊκό σήμα. Νομίζω ότι όπως είπε η συγγήτρια και άλλοι ομιλητές υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Ο αριθμός παραδείγματος αυτών των χώρων είναι σημαντικό. Αν έχουμε ένα σταθερό αριθμό αναχώρες μέλους, μέλου, μπορούμε να θίξουμε ορισμένε χώρες, να τις ε, ε, τι αδικήσουμε σε κάποιο βαθμό. Επίση, ο δημοκρατικό έλεγχο είναι σημαντικό, όχι γιατί είναι εγγύηση ποιότητα, αλλά είναι εγγύηση συμμετοχή των πολιτών και ελέγχου από την πλευρά των πολιτών. Από αυτή την άποψη, εγώ νομίζω θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει στην Επιτροπή μα μια έστω συμβουλευτικού χαρακτήρα συζήτηση επί τη βάση της προτάσεως των εμπειρογνωμόνων. Εμείς δηλαδή δεν θα περνάμε απόφαση, αλλά θα συμμετείχαμε σε αυτή τη συζήτηση, να μπορεί να γίνει μια συζήτηση <clears throat> μέσα στο κοινοβουλευτικό χώρο Έχουμε τώρα πάνω από τέσσερις πολιτικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά, αρκετό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο τέσσερις εκπροσώπους, γιατί αυτό θα εκπροσωπεί την πολυμορφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα επίσης να σκεφτούμε και λίγο μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας για μια σειρά θεμάτων όπως αυτά που ανέφερε και η συγγήτρια στην αρχή της παρεμβασής της λέει αν θα πρέπει αυτό το σχέδιο να παραμείνει μόνο μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα ή αν θα είναι και επέκεινα των ευρωπαϊκών σύνορων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είναι μονάχα ένα θεωρητικού χαρακτήρα ερώτημα. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για το παρελθόν αλλά και για το μέλλον. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει εστραμμένη προς τα μέσα προσπαθώντας να βρει μια ταυτότητα που ίσως είναι και μυθική μια κοινή ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλουμε. Ένας Πορτογάλος όπως εγώ δεν μπορεί να έχει πιο κοινή κουλτούρα με ένα Εστονό από ότι με ένα Βραζιλιανό ή με ένα από το πράσινο ακροτήριο. Αυτό το οποίο λοιπόν για μένα είναι σημαντικό, βλέπω εδώ τον κατάλογο των πολιτιστικών χώρων που έχουν αυτή την ετικέτα στη χώρα μου. Είναι μοναστήρια, βιβλιοθήκες, καθεδρικοί ναοί, ηλική δηλαδή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά έχουμε και άειλη ε, πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι η με ενα απο το πρασινο ακροτηριο αυτο το οποιο λοιπον για μενα ειναι σημαντικο βλεπω εδω τον καταλογο των πολιτιστικων χωρων που εχουν αυτη την ετικετα στη χωρα μου ειναι μοναστηρια βιβλιοθηκες καθεδρικοι ναοι ειδικη δηλαδη πολιτιστικη κληρονομια αλλα εχουμε και αειλη πολιτιστικη κληρονομια οπως ειναι η καταργηση τη θανατική ποινή. Ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κατήργησε τη θανατική ποινή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάθε χρόνο, κάθε μήνα σχεδόν υπάρχει μία συζήτηση στην Ολομέλεια του Στρασβούργου για τη θανατική ποινή εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά. επόμενο, δεν είναι κάτι, δεν είναι μια ετικέτα, ένα σήμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάργηση τη θανατική ποινή είναι ευρωπαϊκή κληρονομιά, όχι, είναι μια συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια κουλτούρα. Δεν λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε τους τίτλους για αυτό το σήμα, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε τη συζήτηση μεταξύ άλλων και στο θέμα αυτό για να δούμε τι κάνουμε με τα θέματα που είναι ευρωπαϊκή συνεισφορά στην παγκόσμια κουλτούρα και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την αναζήτηση μια μυθικής κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ευχαριστώ πολύ. Σα παρακαλώ να σκεφτείτε και το χρόνο. Είναι 6 και 5. Θέλουμε να ακούσουμε και την Κομισιόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάρετε την ε, την θέση μου γιατί θα πρέπει να φύγω για μια στιγμή. Κυρία Κέλλες. Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση. Μέσα από αυτή την πρόταση εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα ήθελα να σας θέσω εδώ ορισμένες προτάσεις αυτό το ευρωπαϊκό σήμα ή αυτός ο τίτλος. Θα πρέπει να αφορά το παρελθόν, αλλά θα πρέπει να είναι και ένα μήνυμα προς το, μένος, προς το μέλος. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό τίτλο για αυτό το σήμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τον τίτλο, θα πρέπει να αναφερόμαστε σε πολιτιστικούς χώρους και μνημεία αλλά επίσης υπάρχουν και άλλες αξίες κοινέ στην Ευρώπη που είναι άειλου χαρακτήρα, που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και είναι επομένως σημαντικό μέσα στα πλαίσια της, ε, των προδιαγραφών για αυτό το σήμα να έχουμε μια σαφή διατύπωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας πολιτιστικός χώρος και μια άειλη συμβολική αρχή. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις. Θα υπάρξει μια προεπιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να έχουν ενιαία κριτήρια για την επιλογή και την προκήρυξη αυτής της, αυτού του Ευρωπαϊκού Σήματος και ελπίζω ότι αυτός ο τίτλος θα μπορέσει να, να γίνει γνωστός και να προσελκύσει και ενδιαφέρον. Τέλος, κάτι το οποίο εγώ θέλω να προτείνω να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο από αυτούς τους τόπους. Αν έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αξίες θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα δίκτυο όλη αυτή η δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λέει κυρία Ράνερ για όλες αυτές τις σχέσεις οι σκέψει αυτέ των συναδέλφων δείξαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω. έχουμε ένα καλύτερο, ένα πιο εστιασμένο προφίλ για την απονομή αυτού του ευρωπαϊκού σήματο. Τι σημαίνει αυτό το σήμα και γιατί το δίνουμε. Η πόλη από την οποία προέρχομαι είχε τον τίτλο του πολιτιστικής Πρωτεύουσα το 2003. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρετε τι σημαίνει αυτό για ένα κράτο μέλο, πόσο ενθουσιάζει το, τους πολίτες μιας ε, πόλης και πόσο ενδιαφέρον δημιουργεί. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σήματα, τα ευρωπαϊκά σήματα, για να προωθήσουμε μια αντίστοιχη διαδικασία στι χώρε μα. Για τα κριτήρια τώρα μα έχει αφήσει πάρα πολλέ δυνατότητε η Κομισιόν. Εμεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία που έχουμε για να καταλήξουμε σε μια πρόταση εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι χώροι ακόμα που έχουν αυτό το σήμα και οι χώροι διακρατικοί όπως ελέγχθη μπορούν να έχουν ενδιαφέρον, αλλά θα ήταν καλό να ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ίσως η γραμματεία, θα ήθελα να ζητήσω από τη γραμματεία να μας πει τι έχει γίνει για τις περιπτώσεις απονομής μέχρι στιγμής σήματος. Κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια Παλιαδέλη γιατί έθεσε τα ζήτηματα κλειδιά για ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό όπως φάνηκε και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι το πέρασμα από μια διακυβερνητική απόφαση που βασίζεται την εθελοντική διάθεση των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μεγάλη ευαισθησία στην επιλογή. Αυτό πρέπει όλοι να το συνειδητοποιούμε πέρα από το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι δύο πτυχές πρέπει να υπογραμμίσουμε. Πρώτον, θα ήταν ενδιαφέρον ίσως να προβλέψουμε ότι τα κράτη-μέλη που επιλέγουν αυτούς τους χώρους ε, ήδη θα πρέπει να ε, λαμβάνουν υπόψη τους τους πολίτες, ε, τις επιστημονικές ενώσεις, τις ενώσεις των πολιτών, μιας και πρόκειται για μια ευρωπαϊκή διαδικασία που έτσι θα ενισχυθεί. Η προεπιλογή από τα κράτη-μέλη και μετά μια επιτροπή, μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά η ε, Κομισιόν. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Ε, δεν θα ήθελα η προεπιλογή από τα κράτη-μέλη εν τέλει να εγκαταλείπεται τελείως. Το κείμενο μας λέει ότι αντίθετα με τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης ή τις περιοχές εκείνες που έχουν κάποιους άλλους χαρακτηρισμούς, η προστιθέμενη αξία αυτού του σήματος θα είναι η βράβευση όχι τόσο ενό ιστορικού μνημείου, αρχιτεκτονικού μνημείου ή καλλιτεχνικού μνημείου, αλλά το γεγονό ότι, εκπροσω... ότι αντιπροσωπεύει συμβολικά την ιστορία, την κουλτούρα αλλά και την ευρωπαϊκή διαδικασία. Παράδειγμα, σε μερικέ χώρε, στη δική μου για παράδειγμα, μεταξύ των μνημείων είναι ε, τα σπίτια όπου γεννήθηκαν ε, οι, τα ιδρυτικά μέλη της Ευρώπης. Αυτό έχει μια συμβολική αξία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ε, θα ήταν επίσης ενδιαφέρον ε, να δούμε τι αντιπροσωπεύουν οι χώροι αυτοί στον υπόλοιπο κόσμο, πώς εκπροσωπούν την ιδιαιτερότητα της Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο αυτό το ειδικό σήμα, να το διαφοροποιήσουμε από το αρχιτεκτονικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα άλλων σημάτων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα να μην ε, ε, χορηγούμε το σήμα αυτόματα, έτσι δύο το χρόνο σε κάθε κράτος μέλος, αλλά πραγματικά να υπάρχει μια ουσιαστική εξέταση της επιλογής που έκανε το, κάθε, το κράτος μέλος. Ε, κάποιος ανέφερε ένα δίκτυο τέτοιων χώρων ή τη διακρατική πτυχή. Κάθε τέσσερα χρόνια θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος και να αφαιρείται το σήμα ενδεχομένως εάν δεν γίνεται σωστή διαχείριση, αν δεν προβάλλεται σωστά ο χώρος αυτός. Λοιπόν, το σήμα αυτό δεν είναι κάτι που χαρίζεται μία φορά και τελειώνει, δεν είναι μια δωρεά ε, και δεν πρέπει και πρέπει να ερμηνεύεται επίσης και ως κάτι που εκφράζει συναισθηματικά τους λαούς της Ευρώπης. Σάκε και ο κύριος και μετά η Ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια για την αναλυτική και εξαντλητική περιγραφή των προκλήσεων. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει εστίαση της προσοχής στην ε, παιδεία και στην ε, εκπαίδευση. Όπως είπαν πολλοί ομιλητές, ίσως η στόχοι μας να είναι κοινή, αλλά η οδός προς την εκτέλεση αυτού του, αυτής της έκθεσης μπορεί να διαφέρουν. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα μας. Επίσης δεν θέλουμε να δημιουργηθεί υπερβολική και τι γραφειοκρατία, ιδίω με τον περιορισμένο μα προπολογισμό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίση τη σημασία μια προσέγγιση από κάτω προ τα επάνω. Θέλουμε να έχουμε τον αντίλογο των πολιτών, τη γνώμη των πολιτών, γιατί στο κάτω-κάτω είναι ένα από του στόχου του προγράμματο αυτού. Μερικά από τα στοιχεία που εθίγησαν στη συζήτηση αυτή μου θύμισε ε, τη συζήτηση που είχαμε για το ευρωπαϊκό Έτο, ε, για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, για την ψηφιοποίησή τη. Θα πρέπει να δούμε πώ θα συμμετάσχουν οι πολίτε και πώ θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα, το διαδίκτυο και όλα τα άλλα ψηφιακά μέσα για να διαδώσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και να ενισχύσουμε την αλληλεπίδραση των Ευρωπαίων πολιτών μεταξύ τους, πολιτών που προέρχονται ίσως από διαφορετικές χώρες, αλλά και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου αν δούμε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον που δημιουργεί το διαδίκτυο, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορούν, μπορούμε να φέρουμε και ανθρώπους εκτός της Ευρώπης να γνωρίσουν αυτή την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Το πρόγραμμα αυτό πιστεύω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια καλύτερη κατανόηση για το τι είναι η Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην το κάνουμε άλλο ένα αδιαφανές, γραφειοκρατικό, πανάκριβο και μάλλον όχι και πολύ σημαντικό εργαλείο. Γιατί και αυτό θα επιδίνωνε την εικόνα που έχει ο κόσμος για την Ευρώπη. Νομίζω πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να είναι αυτό ένα εύχριστο πράγμα, ένα πολύ θετικό πρόγραμμα ένα εύχριστο και θετικό πρόγραμμα και πραγματικά αναμένουμε με ευχαρίστησή μας να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια για να το πετύχουμε αυτό. Ο κύριος Εσκούρια και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ε, ήδη υπόθηκαν πολλά και ίσως η ουσία είναι η εξής. Ε, με ενδιαφέρον άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μας έδωσε μια ωραία και σημαντική και φάνταστη ιδέα την ευρωπαϊκή, που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ταυτότητα και είναι ίσως μια κρίσιμη ιστορική στιγμή και μας έχει δώσει και το γενικό σχηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εργαστούμε. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει φυσικά να εκφράσουμε τη γνώμη μας με μεγάλη σαφήνεια. Πιστεύω λοιπόν ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει στο εσωτερικό όλων των πολιτικών ομάδων ε, και να αποσταλεί στους εισηγητές ε, της κάθε ομάδας, να αποσταλούν στους κάθε ομάδας όλες οι γνώμες και οι αποχρώσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα περιεχόμενο σε, όλον αυτό, σε όλη αυτή τη συζήτηση για το σήμα. Νομίζω ότι πρέπει να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Αυτό το σήμα μπορεί να αποσυρθεί, ε, μπορεί να αξιολογηθεί, ε, μπορεί να αξιολογείται διαχρονικά τι συμβαίνει με την πάροδο του χρόνου. Ίσως θα μπορούσε κανείς κάθε χρόνο να επανεξετάζει το ζήτημα. Ίσως να μπορούν να γίνονται Ίσως να γίνονται και προτάσεις ε, χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με άλλες ε, να δούμε λίγο τον αριθμό των σημάτων που θα χορηγούνται, να δούμε αν θα πρέπει κάποιες χώρες να έχουν περισσότερες δυνατότητες από άλλες. Αναμένω λοιπόν να ακούσουμε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαναλαμβάνω ότι κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να εμβαθύνει, πρέπει να προβεί σε έναν προβληματισμό για το θέμα αυτό, γιατί έχει ε, συνάδει με, την, με το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σκόρια. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι θα πρέπει και η κυρία Μπράνσον από την Κομισιόν να μας δώσει τη γνώμη της Επιτροπής και στη συνέχεια στη συνέχεια μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος ε, θα λάβει το λόγο και μετά 6,5 με γερμανική ακρίβεια πρέπει να τελειώσουμε. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και βεβαίω ευχαρίστω να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τους ερχόμενους μήνες για να βελτιώσουμε το έγγραφο και να εξασφαλίσουμε ότι συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές ανησυχίες. Θα ήθελα να πω, από μεθοδολογική απόψεως, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή η πρόταση βασίστηκε σε ευρύτατη δημόσια διαβούλευση πάνω από 220 οργανισμοί ε, συμμετείχαν, πολλοί εκ των οποίων ήταν ε, αρκετά ε, αντιπροσωπευτικοί και υπήρξε μάλιστα και δημόσια διαβούλευση και μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου και ακρόαση με τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι χρήσιμο λοιπόν να ξέρουμε και για το ιστορικό Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας το 2008, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα το Νοέμβριο του 2008 που καλούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει το σήμα αυτό και υπό το φως των συζητήσεων που έγιναν τότε προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα συμφέροντα των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να αποσαφηνίσω ορισμένα πράγματα για κάποια από τα βασικά για μας σημεία. Πρώτα απ' όλα, η γεωγραφική εμβέλεια. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί στα 27 κράτη-μέλη για την ώρα. Ένας από τους λόγους είναι η ιδέα και ο στόχος του σήματος να έρθουν πιο κοντά οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχε έντονο αίτημα από πλευρά των κρατών μελών ε, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης ε, το σήμα αυτό να είναι συμπληρωματικό με άλλα, ε, με άλλους, με άλλα βραβεία. Θα είναι μια περίπλοκη διαδικασία βέβαια, 27 εθνικές επιλογές κάθε χρόνο και γι' αυτό ακριβώς προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στην ε, αιτιολογική μας έκθεση εξηγήσαμε ότι όταν θα γίνει η πρώτη ε, αξιολόγηση, σε έξι χρόνια από τη στιγμή που θα αρχίσει ε, να ισχύει, τότε μπορούμε να αναθεωρήσουμε εκ νέου τη γεωγραφική εμβέλεια και να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαν και άλλες χώρες να συμμετέχουν στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί και αναφερόμαστε στις, πόλες, στις ε, χώρες που συμμετέχουν στο πολιτιστικό πρόγραμμα, γιατί ακριβώς ε, η χρηματοδότηση θα προέλθει από εκεί. Αυτά ως διευκρίνηση για τη γεωγραφική εμβέλεια. Τώρα, υπήρχε και ένα ερώτημα για την προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας αυτής σε σχέση με άλλες. Πρώτα απ' όλα, το γεγονός ότι πρέπει να βασίζεται στην ευρωπαϊκή ιστορία, στην κοινή οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο συμβολισμός δηλαδή, δεν είναι θέμα αισθητικής ή ομορφιάς των ε, χώρων. Δεύτερον, κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό στην πρωτοβουλία, είναι ότι αφορά σημαντικά σε σημαντικό βαθμό την εκπαίδευση των νέων κυρίως ε, για την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο θέμα ε, διατήρησης ορισμένων χώρων, συντήρησης τους όπως σε άλλες περιπτώσεις. Και τέλος, ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι σε μεγάλο βαθμό η δικτύωση, που είναι κάτι που επίσης ε, κάποιος από τους βουλευτές ανέφερα. Και ένας από τους βασικούς ρόλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα είναι να ενισχύσει ακριβώς τη δικτύωση για την ε, μετάδοση των, των βέλτιστων πρακτικών και για την καλύτερη επικοινωνία βεβαίως. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία απόδοσης του σήματος βάσει του άρθρου 221. Η απόφαση θα είναι εφαρμοστικό μέτρο και αυτό είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία της ε, πολιτιστικής πρωτεύουσα είναι κατά τη διαφορετική και μάλιστα είναι και πολύ μακροχρόνια, 8 μήνες περίπου. Γνωμοδοτεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο αποφασίζει και είναι πολύ ε, χρονοβόρα διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι η πιο ευέλικτη μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που προέκυψε και από τη διαβούλευση, είναι ότι η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοπιστία της όλης προσπάθειας και το κύρος θα εξαρτάται επίσης από αυτό. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται σε ανεξάρτητη διαδικασία επιλογής. Γι' αυτό προτείνουμε οι εμπειρογνώμονες στο Ευρωπαϊκό Πάνελ να είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Προτείνουμε λοιπόν τα ευρωπαϊκά όργανα να τους ορίσουν. Συνεπώς, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει έναν ρόλο στον ορισμό των ε, εμπειρογνωμόνων του πάνελ. Κάτι ακόμη για τον ορισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι γεγονός ότι είναι αρκετά ρευστός, ε, αφορά ε, την ιστορία, συμπεριλαμβάνει και την άειλη κληρονομιά μερικές φορές μπορεί να έχει σχέση και με κάποιον χώρο βέβαια αυτό. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 αναφέρεται ο ορισμός αυτός. Πρέπει να είναι ε, ε, ε, διασυνοριακό διασυνοριακοί χώροι πρέπει να έχουν ε, ε, παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να έχουν κάποια σχέση με ε, πολύ σημαντικά γεγονότα ή προσωπικότητες, να έχουν σχέση με μεγάλες ε, με μεγάλα επιστημονικά ε, επιτεύγματα, αν έχουν ε, παίξει ρόλο στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη. Και επίσης υπήρξε ένα ερώτημα σε σχέση με τον προϋπολογισμό για την πρωτοβουλία. Είναι μάλλον περιορισμένος, αλλά νομίζουμε ότι είναι αποτελεσματικός, ε, τριετής είναι η περίοδος, 1.350.000 ε, χωρίς ε, τα έξοδα του προσωπικού. Δεν θα υπάρξει επιπλέον ε, προσωπικό στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα χρησιμοποιήσουμε το προσωπικό που έχουμε. Είναι περιορισμένο ο προπολογισμό γιατί αυτό ήταν, ε, ήταν η συνένεση μεταξύ των κρατών μελών τότε. Θέλησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά η πρωτοβουλία, να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο ο ε, προϋπολογισμός ε, και γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε επίσης να μην δίδονται απευθείας στους χώρους οι πόροι. Αυτό να επαφίεται στις ε, εθνικές αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά τον αριθμό τώρα των χωρών ε, θα ήταν δύσκολο να ε, δοθούν οι πόροι κατευθείαν σε όλους αυτούς τους χώρους που θα λάβουν το σήμα. Είναι ένα πολύ περιορισμό, περιορισμένο πρόγραμμα. Είναι 400 εκατομμύρια για 35 χώρες και συνεπώς είναι μάλλον περιορισμένο. Όσον αφορά τώρα το λογότυπο, πιστεύουμε ότι είναι μια καλή ιδέα και έχουμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο γιατί θα είναι πιο ορατή η πρωτοβουλία και θα ε, προκαλέσει και το ενδιαφέρον των ε, νέων. Και υπήρξαν και κάποιε ερωτήσεις όσον αφορά την επιλογή και τον αριθμό των χώρων. Θα ήθελα να πω, ειδικά για τον αριθμό, ότι προτείνουμε κατά τη διάρκεια των ετών επιλογής κάθε κράτος μέλος να προτείνει το πολύ δύο χώρους ε, και να επιλέγεται ένας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγεί οπωσδήποτε ένας, δηλαδή αν κανένας από τους χώρους δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί, ε, να επιλεγεί ένας χώρος, ένας όμως είναι ο μέγιστος. Δηλαδή, αν 27 κράτη-μέλη ε, θέσουν όλα υποψηφιότητα θα είναι το πολύ 54 ε, οι, οι χώροι που θα προταθούν. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια για την προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο, τα κριτήρια θα είναι ίδια με αυτά για το Ευρωπαϊκό Πάνελ Εμπειρογνωμόνων, δηλαδή τα κριτήρια του άρθρου 7. Όσον αφορά την οργάνωση όμω, αφήνουμε μεγάλο περιθώριο ελευθερία στα κράτη-μέλη, ε, σύμφωνα με την αρχή τη επικουρικότητα βεβαίω. Μπορούν να οργανώσουν όπως θέλουν την προεπιλογή τους. Πρέπει μόνο να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται τα κριτήρια και ζητούμε να τηρηθεί η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων. Αφήνουμε όμως την ε, ελευθερία οργάνωση στα κράτη-μέλη. Υπήρχαν επίση ερωτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση και την ε, αφαίρεση του σήματο. Στην πρότασή μας ε, έχουμε την ιδέα των τριών ετών ε, επιλογής. Μετά θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και όταν πια θα χειρονταριστεί το σύστημα θα γίνεται ε, κάθε χρόνο παρακολούθηση. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Πάνελ τα σχετικά στοιχεία, το πάνελ θα τα αξιολογεί, θα προβαίνει σε συστάσεις αν χρειάζεται και αν υπάρχουν προβλήματα θα μπορούσε να ξεκινήσει διάλογος ενδεχομένως με τα κράτη-μέλη και τους συγκεκριμένους χώρους για να εξασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και ότι τα κριτήρια γίνονται σεβαστά. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση στο τέλος της διαδικασίας, αν οι χώροι δεν σέβονται τα κριτήρια, ακόμη και μετά τις ε, συστάσεις, τότε ενδεχομένως ε, να αφαιρεθεί το σήμα. Και η ιδέα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τη σχετική απόφαση βάσει της αξιολόγησης του πάνελ. Όπως ε, θα λάβει και την απόφαση δηλαδή για την απόδοση του σήματος. Θεωρητικά βέβαια δεν, εμποδίζει, δεν εμποδίζεται κανένα χώρο ε, να υποβάλει και πάλι την, ε, να είναι και πάλι υποψήφιος ε, σε μεταγενέστερο στάδιο και ευχαρίστω να απαντήσω ερωτήσει, αν θέλετε. Σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο. Δίνω το λόγο και πάλι στην κυρία Παλιαδέλη. Έχετε το λόγο κυρία Παλιαδέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Επιτροπής για τις διευκρινιστικές συμπληρώσεις αυτά που ε, ε, παρουσίασα με την εισήγησή μου. Χαίρομαι ότι το λογότυπο, ο λογότυπος ε, είναι από τα ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ε, να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι όταν μιλούσα για μνημεία ή για τόπους, βεβαίως εννοούσα ε, και ιδέες και άειλα ε, άειλη πολιτιστική κληρονομιά με, με όλους τους δυνατούς τρόπους. Βεβαίως, μια, ένας τέτοιος τεράστιος ορισμός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στα κριτήρια. Δηλαδή είναι πραγματικά δύσκολο και εδώ θα ήθελα πολύ τη βοήθειά σας για να δούμε με ποιο τρόπο θα διαμορφώσουν τα κριτήρια. Γιατί υπάρχουν διαμορφωμένα στην πρόταση, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόταση ε, είναι κομμάτι μιας διαδικασίας που αφορά στη συναπόφαση. Δηλαδή οδηγεί σε συναπόφαση, που σημαίνει ότι όπου δεν συμφωνούμε θα πρέπει να ξανακουβεδιάσουμε. Έχουμε δηλαδή δύο ή τρεις φορές μέχρι ότου καταλήξουμε σε κοινέ αποφάσεις, προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για ένα τέτοιο σημαντικό ε, θεσμό, όπως αυτός που προτείνεται με την ε, πρόταση αυτή. Για μένα λοιπόν το βασικό είναι ο ορισμός του, του, του σήματος ή μάλλον της πολιτικής κληρονομιάς και τι εκφράζει το σήμα μέσα από αυτό, τα κριτήρια και δυστυχώς και ο προϋπολογισμός. Δεν ξέρω, ο προϋπολογισμός είναι συνάρτηση ως ένα βαθμό και του αριθμού των ε, αποδεκτών του σήματος. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Αν έχουμε 21 χώρες, κάθε, 21, 21 σήματα κάθε χρόνο, πέρα από το ότι πέφτει η, η, η ποιότητα, το κύρος του θεσμού, κάθε χρόνο 21. Σε 10 χρόνια 210. Ε, Δεν ξέρω αν είναι το σωστό, το πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Πέρα λοιπόν από το ότι πέφτει το κύρος του θεσμού, άρα θα πρέπει να δούμε πιο ευέλικτα το ζήτημα των αριθμών των αποδεκτών αυτού του σήματος, θα πρέπει <clears throat> να ε, αποφασίσουμε ως ένα βαθμό και για, ίσως και για περισσότερα σήματα. Είναι δύσκολο όλα αυτά να είναι κομμάτια του ίδιου σήματος. Είναι τεράστιος ο ορισμός, πρέπει να τον ξανασκεφτούμε. Ε, έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη μου τις παρατηρήσεις. Συμφωνώ ιδιαίτερα, θα ήθελα να το δηλώσω παρόλο που δεν είναι εδώ ο συνάδελφος, ότι η πρότασή του, ο κύριος Ταβάρες, <clears throat> ότι η πρότασή του για τον συμβουλευτικό ρόλο της Επιτροπής Πολιτισμού στη λήψη των, της απόφασης της Επιτροπής θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα που έθεσα σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Ως έστω συμβουλευτικός μέσω εκπροσώπων του Κοινοβουλίου που μετέχουν στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Ε, και πραγματικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στα 27 κράτη, ακόμη και αν για τεχνικούς λόγους υπάρχουν επιχειρήματα σαν αυτά που μας είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πιστεύω ότι πρέπει να, πραγματικά να διευρύνουμε το, τους στόχους μας, να βγούμε έξω από τα όρια της Ενωμένης Ευρώπης, να, να παραμείνουμε τουλάχιστον στα όρια της Ευρώπης, αν όχι να ακολουθήσουμε την άποψη του κ. Ταβάρες που έφερε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τη συνεισφορά της Ευρώπης στην παγκόσμια κουλτούρα με αφορμή την κατάργηση της θανατικής ποινής για πρώτη φορά στην Πορτογαλία. Επομένω, είναι ζητήματα για τα οποία θα ξανακουβεντιάσουμε με την Επιτροπή και θα ήμουν ευγνώμων, το email μου είναι εύκολο να το βρείτε, ό,τι ιδέα έχετε ω μέλη τη Επιτροπή, θα ήμουν ευγνώμων να δέχομαι μηνύματα, θα, βοηθήσουν πάρα πολύ στο στήσιμο του σχεδίου τη απόφαση που θα έχετε στα χέρια σα σε ένα περίπου μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Παλιαδέλη, και ο πρόεδρος. Θα εξετάσουμε και πάλι το θέμα αυτό στις 2 Σεπτεμβρίου. Αύριο ξεκινάμε με την συνάντηση των συντονιστών στις 9 και στη συνέχεια στις 9 και 45 η κανονική μας συνεδρίαση. Γεια σας μέχρι αύριο